Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αρχίζει η συνεδρίαση και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καθίσετε στις θέσεις σας. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση και θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω ότι η γραπτή δήλωση για την καταπολέμηση της ε, σκλήρινσης ε, κατά πλάκα στην